και, και το κοινοβούλιο με μια έννοια εκείνο που μας ενδιαφέρει όμως τουλάχιστον είναι τα κονδύλια αυτά να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο και με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Η συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Λάμπερ σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την επιτροπή για τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης το 112 για τη μη εφαρμογή του ψηφίσματος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου του 2011 και του άρθρου 26 της οδηγίας 136 του 2009 ε, εκ των ε, εισηγητών έχω δύο συναδέλφους που θα παρουσιάσουν την προφορική ερώτηση και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να παρακαλέσω τη συνάδελφο φιόνα χολ να πάρει το λόγο για μισή λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ το χρησιμοποίησα το νούμερο αυτό και η βοηθός μου το χρησιμοποίησε. Φαντάζομαι και άλλοι εδώ όταν υπήρχε ανάγκη να το χρησιμοποιήσω χάρηκα που μπορούσα να το χρησιμοποιήσω αλλά 50% των Άγγλων συμπατιωτών μου δεν γνώριζαν τίποτα για το νούμερο αυτό άρα θα πρέπει να κάνουμε κάποια δουλειά για να προωθήσουμε τον αριθμό αυτό κλήσης μπορεί να μας πει η Κομισιόν τι θα κάνει για να πει στα κράτη-μέλη να προωθήσουν το νούμερο. Και κάτι τι άλλο τώρα. Πρόσβαση για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρίες. Εκατομμύρια ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση γιατί είναι κουφοί, είναι βαρύκοοι ή έχουν άλλες ειδικέ ανάγκες. Άρα χάνουν ένα δικαίωμα που έχουν για την, ε, για την υπηρεσία αυτή. Στην πρόσφατη δήλωση του 35-2011 ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί πρόσβαση για τους ανάπηρους πολίτες και ειδικά η Κοφή και η Βαρύκοη δεν ελέγχει διότι ελέγχθη ότι οι και οι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή παρά μόνο ε, στην επόμενη γενιά. Θα ήταν όμως καλό να ε, φροντίσουμε ε, να υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Στο ψήφισμα της 5ης Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε κονδύλια για να χρηματοδοτήσει αποκτήσει ακριβώς ε, νέες τεχνολογίες για την περίπτωση αυτή, για τη χρησιμοποίηση του αριθμού μέσω ίντερνετ ε, και για να αναπτυχθεί το σύστημα νέας γενιάς του συστήματος αυτού. Ε, οι κανονισμοί επίσης που σχετίζονται με το 112 μέσο διαδικτύου και με τους παρέχοντες υπηρεσία εκεί ε, στο διαδίκτυο, ε, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν γρήγορα και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 112 είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Αναμέναμε να αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα στα διάφορα μέρη της Ευρώπης. Ωστόσο η εφαρμογή ε, δυστυχώς έχει καθυστερήσει και η ερώτηση είναι ε, θέλουμε ε, να ξέρουμε γιατί συνέβη αυτή η καθυστέρηση. Μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την ασφάλεια των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα σε περίπτωση κάποιες καταστροφής ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα τους εγγυηθεί την άμεση βοήθεια αξιόπιστα. Όταν ε, χρειάζεται βοήθεια σε επίγουσα ανάγκη, θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να βασιστεί σε ένα αποτελεσματικό σύστημα, ε, τάχη, ε, αποδοτικό, αποτελεσματικό και πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν χρειάζεται επίγουσα βοήθεια, μιλάμε για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο. Το θέμα λοιπόν είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω το 112 και είναι εξίσου σημαντικό οι συμπολίτε μα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορε γλώσσε. Κατανοώ ότι όταν είναι κανεί στη Γαλλία θέλει να έχει πρόσβαση ε, στα γαλλικά και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να εργαζόμαστε με το, σωστά με το 102, να έχουμε τηλεφωνητές που να μπορούν να μιλούν τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά θα πρέπει να προσέξουμε και το γλωσσικό θέμα δηλαδή που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια στα διάφορα κράτη-μέλη χρειάζεται να υπάρχουν υπηρεσίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της συγκεκριμένη ε, χώρας, όπως ας πούμε στη Φιλανδία, στα Σάμι, τα Φιλανδικά και τα Σουηδικά. Εάν ληφθεί λοιπόν υπόψη και το γλωσσικό θέμα, θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επίσης, πιο αποτελεσματική ενημέρωση, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει την ύπαρξη του αριθμού αυτού. Έρευνες δείχνουν ότι πολύ λίγος κόσμος το γνωρίζει ακόμα. Γι' αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί η ενημέρωση του κόσμου. Ο Επίτροπος το λόγο, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν σκοπεύει βεβαίως να διασφαλίσει καλύτερη ενημέρωση και εφαρμογή του αριθμού 112 στα κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ έχει λάβει κάποια μέτρα για τα ζητήματα που ανέφερε το Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε πως η Κομισιόν πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για να προωθήσουν το 112. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο Κάλλας ζητήσαμε από τις εταιρείε μεταφορών να ενταχθούν σε μια καμπάνια για να ενημερώνουν τους πελάτες τους από χώρα σε χώρα. Και τώρα κάναμε το ίδιο και με τους tour operators στην Ελλάδα μαζί με τις αρχές θα κάνουμε μια καμπάνια με βίντεο και το ίδιο θα γίνει και σε άλλα κράτη-μέλη. Και βεβαίως ε, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για πρόσβαση στις υπηρεσίες άμεσης ανάγκης και θα πρέπει οι αρχές ε, να δώσουν κάποια, να ορίσουν κάποια κριτήρια για την κατανομή των ε, τηλεφωνημάτων και βεβαίως μην ξεχνάμε πώς η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να υπάρξει ακριβώς μία συναντήληψη για τα κριτήρια αυτά. Πέρσι δε οι υπηρεσίες της ε, Νέλη μαζί με τα κράτη-μέλη ανέπτυξαν κάποιους δείκτες ε, κλειδιά για να διευκολυνθεί η σύγκριση των δεδομένων της εφαρμογής του 112. Με βάση λοιπόν το πιλωτικό αυτό έργο θα ανασχεδιάσουμε τις αναφορές οι οποίες δίνονται κάθε χρόνο και θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα για το πώς ε, λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές στα κράτη-μέλη. Επίσης θα υπάρξει μια αξιολόγηση της λειτουργίας των υπηρεσιών και βεβαίω η ανάπτυξη ενός αντίστροφου τέτοιου συστήματος είναι ένα ζήτημα που είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όσον αφορά δε τις βέλτιστες πρακτικές υπάρχει και η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Υπάρχει επίσης ε, ένα πιλωτικό έργο όσον αφορά τη βελτιωμένη προσβασιμότητα σε πέντε κράτη-μέλη που έχει επιδείξει την δυνατότητα συνομιλιών που θα συμπεριλαμβάνουν φωνή, κείμενο και βίντεο και απαιτείται βεβαίως περαιτέρω τυποποίηση. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Σβάμπ για το ΕΛΚ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδέλφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έκαναν αυτή την ερώτηση, αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι Ράπτη και Τούν πριν από λίγους ημίνες στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε, κύριε Επιτροπέ, για την ψηφιακή εσωτερική αγορά, τις δυσκολίες που έχουμε για να ολοκληρωθεί αυτή και το βλέπουμε αυτό στον αριθμό 112 που παραδείγματο χάρη όταν πάει κανείς διακοπές θα τον διευκολύνει ε, να ε, ξέρει που πρέπει να πάρει τηλέφωνο εάν χρειάζεται βοήθεια. Γι' αυτό θεωρώ πως το παράδειγμα του αριθμού 112 που δεν λειτουργεί ακόμα σε όλα τα κράτη-μέλη όπως ε, θα έπρεπε ε, πως πρέπει να αυξήσουμε την πίεση. Γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς κύριε Επίτροπε έτσι ώστε να πέσουν ακριβώς αυτά, αυτοί οι φραγμοί που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά και να υπενθυμίσω και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τάκουλα πρέπει επίσης να υπάρξει η προσαρμογή στην ε, γλώσσα του καλούντος. Γιατί ε, αυτό ισχύει βεβαίως σε αυτή τη στιγμή μόνο για όσους μιλάνε τη γλώσσα της κάθε χώρας. Δεν είναι αυτό ικανοποιητικό. Νομίζω το e-call ε, που υπάρχει και στα γιοταχή νομίζω πρέπει να επεκταθεί. Σας ευχαριστώ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 Ο αριθμό ε, έκτακτη ανάγκης 112 είναι μια από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίε. Είναι δωρεάν κλίση ε, για οποιονδήποτε ε, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωση, οπουδήποτε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωση, Είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και παρά τα πλονεκτήματα που προσφέρει, η γνώση και η χρήση του είναι ακόμα ελλειπής. Ε, πρέπει να εφαρμοστεί ε, ε, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο. Ε, το άρθρο 26 της οδηγίας εγγυάται την ίση πρόσβαση στους, στους ανάπηρους αλλά και δίνει τη δυνατότητα μόνο σε 13 κράτη-μέλη. Πολλοί πολίτες δηλαδή δεν μπορούν να έχουν αυτή την επιλογή. Επίσης σε περίπτωση αυτοκινητιστικού. θα έπρεπε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έπρεπε να είναι επιχειρησιακό στη 2012. Ε, ε, αλλά υπάρχει καθυστέρηση. Θέλω να γνωρίζω πώς σκοπεύει να προωθήσει η Κομισιόν την ε, την υποδομή που χρειάζεται ώστε να προωθηθεί η χρήση του 112. Ελευθέρω. Yes, uh, thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ηνωμένου Βασιλείου γνωρίζουν ότι όπου και να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του 112 είναι ένα από τα πολύ συγκεκριμένα εργαλεία που προσφέρει η Ευρώπη στους πολίτες της και δίνει μια ασφάλεια, μπορεί να σώσει ζωές σε ορισμένες, περιστάσεις. Αλλά δυστυχώς ο Ευρωπαίος πολίτης δεν γνωρίζει την υπηρεσία αυτή. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και προέρχεται από τα κράτη-μέλη και την ε, εφαρμογή του 12 Του 112 ε, ε, έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη για παράβαση από 15 κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ φοβερό το ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν προωθήσει ε, κάτι αντίστοιχο με την ηλεκτρονική κλίση, το e-call. Εγκαθίσταται σε αυτοκίνητα. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και με το 112. Κάτι θα μπορούσε να ε, έχει ήδη γίνει και ε, ξέρουμε ότι στο μέλλον θα είναι υποχρεωτικό να έχουν το e-call τα αυτοκίνητα οπότε θα μπορούσε να συνδεθεί με το 112 από εκεί και πέρα τι γίνεται άμα θέλει κάποιος να πάρει από το κινητό του το 112 Λοιπόν, τα κράτη-μέλη έχουν φτιάξει τα συστήματά τους ε, έτσι ούτως ώστε να μπορούν να δεχθούν τα 112 και τις ηλεκτρονικές κλήσεις από τα αυτοκίνητα και η Κομισιόν τι θα κάνει για την κάλυψη όλου του ευρωπαϊκού χώρου από, του, από κινητά τηλέφωνα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κενά. Ε, κάτι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένες μέρη δεν υπάρχει κάλυψη. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Η κύριε Ιζαμπέλ Ντουγόν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω πώ σε ορισμένου τομεί προχωράμε ταχύτατα. Ασκούμε τη μέγιστη πίεση, αν δούμε ας πούμε τις ε, ε, τον προπολογισμό ή άλλα θέματα όπου τα κράτη-μέλη δείχνουν μεγάλη ικανότητα και αποτελεσματικότητα για την εφαρμογή ενό μέτρου. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Το 112 αυτή τη στιγμή δηλαδή το γνωρίζει ένα στου τέσσερι Ευρωπαίου πολίτε. Μα λέτε διάφορου δρόμου διάφορο... που έχει ακολουθήσει η Κομισιόν. Θέλω ωστόσο διευκρινήσει για το πώ ακριβώ ε, οριζόντια θα πρέπει να συνοηθούν οι διάφορε υπηρεσίε τη Κομισιόν προχωρήσουν τα πράγματα. Αναφέρθηκαν και κάποια παραδείγματα, αλλά να μα πείτε επίση πού είναι το πρόβλημα στα κράτη-μέλη. Πείτε μας το για να μπορέσουμε κι εμεί ε, να πούμε στα κράτη-μέλη μα την ανάγκη να προχωρήσουμε για πράγματα τα οποία είναι προβληματικά. Ε, επίσης, είναι πολύ σημαντικό την ε, στιγμή που η τεχνολογία στον 21ο ε, αιώνα όπου τα πράγματα είναι όπως είναι η τεχνολογία είναι αυτή που είναι να είμαστε σε αυτή την κατάσταση δεν είναι αποδεκτό πρέπει πραγματικά να πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε επίπεδο της Κομισιόν αλλά και κρατών μελών για να έχουμε από γρήγορα αποτελέσματα πραγματικά ε, ε, να λειτουργήσει το σύστημα αυτό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατά κάποιον τρόπο είναι απογοητευτικό το ότι πάλι το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει πίεση στην Κομισιόν για αυτό το ζήτημα. Και οφείλω να αναγνωρίσω τους συναδέλφους που εργάστηκαν επί του θέματος, αλλά μια που ήμουν ο εισηγητής της έκθεσης που πέρασε το 2002 και ζητούσε την πλήρη εφαρμογή του 112, και πληροφορίες για την κατανομή της κλίσης και υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για την καθολική παροχή υπηρεσίας το 2009 και επιπλέον υπάρχει η έκθεση του κυρίου Σβάμπ για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν έχει τάση η στιγμή να αναλάβει η Κομισιόν τις ευθύνες της. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε κάτι στο οποίο δεν αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι και αφορά τα δεδομένα θέσεις του ε, καλούντος και έτσι βοηθάμε τον κόσμο. Είναι πράγματι ζωτική σημασία για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής κλήσης που ανέφερε ο κ. Μπένιαν. Αυτή η διάταξη υπήρχε στην έκθεση του 2002 και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν κοινέ τεχνικές προδιαγραφές για γρήγορες και ακριβείς πληροφορίες. Ακόμα δεν το έχουν κάνει, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζουμε πως τεχνολογία υπάρχει. Οπότε επιμένω πως η Κομισιόν πρέπει να κινητοποιηθεί επιτέλους για αυτό το ζήτημα και το των δυνατόν και να μην δεχτούμε άλλες απαραδέκτες καθυστερήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Ευχαριστώ. Πρέπει βεβαίω να προωθήσουμε το 112 όπω του αξίζει και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Επιτροπό τι άλλο μπορεί να γίνει. Γιατί παρά το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα το 2011, ψήφισμα το οποίο ζητούσε μεγαλύτερη προώθηση του αριθμού, τα αποτελέσματα δεν ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά όπως ακούσατε. Είναι λυπηρό το ότι σε μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πάνω από 25% των ερωτώμενων μπορούσαν να αναγνωρίσουν ποιος είναι ο αριθμός τον οποίο μπορούν να καλούν σε οποιαδήποτε χώρα. Στη χώρα μου 14% των ερωτώμενων μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για τον αριθμό παρά το ότι υπήρχε προσδοκία πως οι χώρες θα ενημέρωναν τον πληθυσμό. Μιλάμε για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη, αλλά και πολλέ άλλε χώρες δεν τα πάνε πολύ καλύτερα. Καθώ λοιπόν πλησιάζουν οι διακοπές και εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό, νέοι και γέροι, πρέπει να θυμόμαστε τη σημασία του 112 που προφανώς χρειάζεται περισσότερη διαφήμιση. Εγώ Άρχισα να το προωθώ προσφάτω, για να παίξω και εγώ τον δικό μου ρόλο, αλλά συμφωνώ και με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την κυρία Χολ για την σημασία της ίσης πρόσβασης του 112 για όσους είναι βαρύκοοι οικοφοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Προς τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές, πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στην συνάδελφο Τούν για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα δεδομένα είναι αρκετά άσχημα όσον αφορά τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Ε, ε, πολλοί κόσμος χάνει τη ζωή του κάθε χρόνο και 105.000 περίπου μένουν άπειροι. Τα αυτοκινητιστικά είναι η ένατη αιτία θανάτου, ήταν μάλλον η ένατη αιτία θανάτου το 2004 και μέχρι το 2020 ε, εάν έχουμε τέτοια πρόοδο θα φτάσει να γίνει τρίτη αιτία. Κυρίως υπό το φως των επικείμενων ε, διακοπών ε, πρέπει να σκεφτούμε ότι το 112 μπορεί να σώσει πολλές ζωές και συμφωνώ με τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και χαίρομαι όσον αφορά το e-call. Το e-call ναι, μπορεί να ε, σώσει 3.000 το άνθρωπους του χρόνο, αλλά δεν θα είναι αποτελεσματικό αν δεν θα λειτουργήσει πρώτα το 112. Θα πρέπει να είναι γνωστό, να, μάλλον να καλύπτεται το σύνολο του ευρωπαϊκού ε, χώρου, της ευρωπαϊκής επικράτησης. Ευχαριστώ. Όλοι οι συνάδελφοι συμφωνούν. Η διαπίστωση είναι ότι έχει τελματώσει η γνώση του 112 στους τέσσερις ε, πολίτες το ξέρουν. Τα κριτήρια εντοπισμού δεν έχουν καθοριστεί. Η λειτουργία του συστήματος είναι ατελής σε πολλά κρατημέλη. Αντιθέτως για το e-call το οποίο στηρίζει η Κομισιόν τα όλα ήταν πιο απλά και πιο γρήγορα. Οι βουλευτές κλήθηκαν στις ομάδες εργασίας. Αυτό δεν συνέβη με το 112 γιατί συχνά μας αρνήθηκαν την πρόσβαση σε συνεδριάσει που διοργανώνονταν στις Βρυξέλλες ενώ εμείς ήμασταν στο Στρασβούργο. Γι' αυτό και έχω τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, να ρωτήσω αν η Κομισιόν είχε κάτι να κρύψει όσον αφορά τα 112 δεδομένε τη μικρότερη πρόοδου που έχουμε κάνει. Ε, Ο προπολογισμό ο ετήσιο επίση είναι μικρότερο, αλλά και οι δομέ που έχετε φτιάξει για να ευνοήσετε τη συνεργασία ανάμεσα στι διάφορε υπηρεσίε τη Κομισιόν για αυτό το θέμα. Και τέλο, ο προπολογισμό που έχετε κάθε ε, χρόνο για την προώθηση του 112 είναι ένα θέμα ε, εμβληματικό, ένα σημαντικό μήνυμα για του πολίτε ε, αυτή τη ραγμένη περίοδου. Αυτά είναι θέματα που θα έπρεπε να βιαστούμε για να δείξουμε στου Ευρωπαίου, στου πολίτε, ότι η Ευρώπη οποίο είναι ένα συν, ιδιαίτερα όταν δυσκολεύονται, όπως ας πούμε στις περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης. Ε, ελπίζω λοιπόν πώς θα μας δώσετε τις εθαρρυντικές πληροφορίες ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, το άρθρο 26.3 της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσία λέει ότι θα πρέπει το νούμερο 112 να υπάρχει σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο και να εφαρμόζεται σωστά οι πολίτες ε, είναι, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ε, να έχουν αυτοπεποίθηση όταν τηλεφωνούν στο 112 γιατί μπορεί να είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Πρέπει να ε, έχουμε καλή ποιότητα υπηρεσίας επίσης για το 112. Άρα χρειαζόμαστε δεδομένα. Ερώτηση. Οι Κομισιόν, τα κράτη-μέλη έχουν τέτοιου είδους δεδομένα για το πώς αντιμετωπίζονται οι κλήσεις στο 112 και στα εθνικά νούμερα έκτακτης ανάγκης και η σύγκριση μεταξύ του 112 και των εθνικών αριθμών κλίση έκτασης ανάγκης ποια η, ε, η σύγκριση αυτή τι μας δίνει πρέπει να ή κάνουμε μια σύγκριση αντικειμενική και να δούμε τα στοιχεία. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν, ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν εσείς ζήσατε ποτέ μια κατάσταση σοκ μετά από ένα γεγονός που απείλησε τη ζωή σας ή μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να σας έρθουν στο μυαλό κάποια νούμερα επίγουσας ανάγκες. Και όταν φεύγετε και πάτε διακοπές στη Νότια Γαλλία, στη Φινλανδία ή σε μια άλλη χώρα θα πρέπει να, σκε... να έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε το ίδιο νούμερο. Όλοι θα έπρεπε να γνωρίζουν ένα ενιαίο νούμερο, διότι ε, για αυτούς όλους τους λόγους είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αριθμός 112 και το e είναι πολύ σημαντικό σε ένα μνημόνιο συνεννόηση τα κράτη-μέλη συμφώνησαν για το e ε, αλλά πρέπει να λειτουργήσει το 112 πρώτα Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο τον έφερε αυτό σε ένα ψήφισμά του ότι το e-call στα αυτοκίνητα εξαρτάται από το 112. Πρέπει λοιπόν όλοι να αγωνιστούμε ούτω ώστε να εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο το 112. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξοπλίσουν τα τηλεφωνικά κέντρα τους με hardware και με software που να αντιμετωπίζει το Συγχωρείς, κλείσει 112. Η Κομισιόν τι κάνει. Ο συνάδελφος Σέρτου Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει ότι χρειάζεται ένα ενιαίο νούμερο ε, έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη. Όμως αυτά τα είπαμε ήδη τη δεκαετία του 90. Τώρα 25% μόνο των πολιτών γνωρίζουν το 112. Στην Ιταλία 5% μονάχα και στην Πολωνία 50%. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προωθήσουμε το 112 και τη δυνατότητα εντοπισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα του καλούντος αλλά και στο εξωτερικό να υπάρχει ε, σύστημα εντοπισμού αυτόματο και όπως ελέγχθη ήδη είναι, αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα το συνδέσουμε αργότερα με το e-call Ακούσα ότι θα γίνει πρόταση μέχρι το τέλος 2000 μέχρι το τέλος του 2014 για το τι θα γίνει ακριβώς ερώτηση κομισιόν τι θα κάνει μέχρι το τέλος του 14. θα κάνει κάτι τι. Συνάδελφος Γκάλ Πέλτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που δώσατε και για τη σημασία που αποδίδεται στο ζήτημα αυτό, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, ότι πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια συνεχής αξιολόγηση για να δούμε το εάν αυτό το σύστημα που μπορεί να σώσει ζωές λειτουργεί ικανοποιητικά. Να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Το 2006 εισήχθη αυτός ο αριθμός στην Ουγγαρία και έχουμε εξοδέψει μέχρι το 2012 19 εκατομμύρια ευρώ για να προωθήσουμε το σύστημα, να καταργήσουμε τους προηγούμενους αριθμούς και να εισαχθεί ο νέος ε, αριθμός στη χώρα μου. Πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω αυτοί οι στόχοι. Συμφωνώ και με τον κύριο Χάρμπορ γιατί στον 21ο αιώνα ε, ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα σύστημα χωρίς μια κοινή βάση πληροφορικής, ένα σύστημα ε, αναζήτησης δεδομένων και κατανομής των κλήσεων. Επίσης πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση για όλους τους πολίτες και για αυτούς οι οποίοι έχουν αναπηρίες γιατί αντιμετωπίζουν ε, αυξημένες ε, δυσκολίες. Η εμπειρία μου δεν είναι πάρα πολύ καλή ως προς αυτό. Σε κάποια κράτη-μέλη προσπάθησα να τηλεφωνήσω στο νούμερο και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης ε, και ανταπόκρισης. Πρέπει να ενοποιηθεί λοιπόν το σύστημα για να είναι προσβάσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω πως η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, οι στόχοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όλοι λένε το ίδιο, όλοι οι ευρωβουλευτές ζητάνε από την Κομισιόν να επεκτείνει την διαθεσιμότητα του συστήματος, ε, την ενημέρωση για το σύστημα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Όχι κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά αμέσως πρέπει να λάβουμε μέτρα. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και αναμένουμε βεβαίω καθοδήγηση από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Το 112 είναι μια θετική κατάκτηση για μπορεί ο καθένας να τηλεφωνήσει δωρεάν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να είναι μια επιτυχημένη υπόθεση, αλλά δυστυχώς όπως ακούσατε δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες και είναι και σύμβολο νομίζω της ανικανότητας ε, της Ευρώπης να λύσει προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα κοινό τέτοιο νούμερο που να λειτουργεί. Πραγματικά θα μπορούσε να είναι σύμβολο για το ότι κάνουμε κάτι από κοινού. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους να το λειτουργήσουμε το σύστημα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι από εμά δεν αντιμετώπισαν ποτέ μια επίγουσα κατάσταση σε χώρα του εξωτερικού και να αναρωτιέται τι νούμερο πρέπει να, κάνει, να καλέσει. Το 112 είναι η απάντηση σε τέτοιες καταστάσεις. από την Ισπανία στη Φιλανδία, την Πολωνία, την Τσεχία, το νούμερο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλέσει βοήθεια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Είναι δωρεάν και αυτό είναι πολύ ε, μεγάλο πλεονέκτημα όταν ξέρουμε ποια είναι τα κόστη. Το 112 λοιπόν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που διευκολύνει την, την ζωή των συμπολιτών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, ε, ενημερώσουμε για αυτή την χρήσιμη πρωτοβουλία για τους πολίτες. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τους ευρωϊπαλλήλους που εργάζονται στο Ισβρυξέλλες και γνωρίζουν τον αριθμό αυτό. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον να δουλέψει η Κομισιόν για μια μεγάλη διαδικασία στρατηγική ενημέρωση για να προσπαθήσει να προωθήσει το 112. Θα πρέπει βέβαια να βελτιωθεί και το νούμερο αυτό. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι δουλεύουν ε, μόνο σε μερικές γλώσσες της Ένωσης είναι ένα μειονέκτημα και μάλιστα θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην αρχή της πολυγλωσσίας που κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κλήσει θα πρέπει να βελτιωθούν για 6 εκατομμύρια κλήσει ετησίω. οι υπηρεσίε επίγουσες βοήθεια χάνουν πολύ χρόνο ενώ παίζονται ανθρώπινε ζωέ δεν υπάρχει χρόνο για χάσιμο είναι πολύ σημαντικό να μην εισάγονται διακρίσει με το 112 και να εξασφαλίζονται, εξασφαλίζεται ότι οι οι κοφάλαλοι επίσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιήσουν αυτό το νούμερο. Στο σύστημα με SMS ας πούμε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κλείσω λέγοντας ότι καλύτερα είμαστε στο Στρασβούργο, ας παραμείνουμε εδώ, είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Jordan. Πρόεδρε, για να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας χρησιμοποιούμε ε, τα social media αλλά τους ρώτησα, εγώ ρώτησα παρόλα αυτά τους πολίτες μου για το αν γνωρίζουν το 112 και μου έκανε εντύπωση που απάντησαν μαζικά ότι γνωρίζουν το νούμερο. Άρα οι πολίτες της Σλοβενίας γνωρίζουν τον αριθμό κλήσεις για έκτακτη ανάγκη και οι εμπειρίες τους ε, κατά την κλίση αυτού του αριθμού είναι καλές. Ζητώ από την Κομισιόν λοιπόν να ε, φτιάξει ένα ε, κείμενο για να δώσει οδηγίες για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε γιατί είναι εφαρμόσιμο τι πρέπει να εφαρμόσουμε μάλλον για να μπορεί να λειτουργήσει καλά το 112. Πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε και τους ανθρώπους με αναπηρίες. Επίσης να φροντίσουμε να καλύψουμε όλες τις γλώσσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τη λειτουργία αυτού του αριθμού υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα μόνο είναι 27% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν πως υπάρχει αυτό το νούμερο παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το τι γίνεται με την πληροφόρηση. Ένα άλλο ανησυχητικό ζήτημα είναι η μέθοδος εντοπισμού του καλούντος. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα των ατόμων με αναπηρίες. Επίσης οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, βλέπουν πως δεν υπάρχει κάλυψη σε περιοχές της υπαίθρου. Ένα άλλο θέμα είναι ο εξοπλισμός των υπηρεσιών ε, ανάγκης. Ε, απαιτείται λοιπόν μια στρατηγική έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός διασυνοριακός και περιφερειακός. Πολύ η συνάδελφος Πρένεργας. Uh, thank you. Um, like other speakers here this morning, um, there is... Όπως και άλλοι εδώ, uh, θα πρέπει πιστεύω να προωθήσουμε το 112 γιατί στην Ιρλανδία δεν ήξεραν να πούμε ποιο νούμερο να πάρουν σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης βέβαια ε, πρέπει να διαδώσουμε αυτό το πολύ απλό και σημαντικό νούμερο επειδή επιπλέον όλο ένα και περισσότεροι νέοι ζουν ε, στην Ευρώπη, παντού στην Ευρώπη ε, για να σπουδάσουν ή για να ζήσουν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και οι, τα, οι ανάπηροι. Ιδιαίτερα στι απομακρυσμένε περιοχέ, στι περιοχέ τη Υπαίθρου, το θέμα είναι σοβαρό. Θέλω ωστόσο να τιμήσω την ε, συνάδελφο Σαρονόβα για την προσπάθεια που ήδη έχει καταβάλει. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, ειδικά για όσους ταξιδεύουν και δεν έχουν ε, συγγενείς ή φίλους ε, με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος ε, σε αυτό τον αριθμό. Και αυτό συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Επίτροπος ε, και καλωσορίζω αυτό το οποίο είπε ότι θα κάνει για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο νούμερο αυτό. Επιπλέον, όπως είπε και η Φιώνα Χολ, πρέπει να διαδώσουμε τις ε, πληροφορίες για να ε, είναι δυνατή η χρήση και από ανθρώπους με αναπηρίες, ειδικά τους ε, κοφούς και όπως είπε και ο κύριος Τάκουλα θα έπρεπε νομίζω και κάποιες γλώσσες όπως τα αγγλικά γαλλικά να ομιλούνται παντού. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το 112 μπορεί να σώσει ζωές, έχουμε όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα, ο κόσμος ταξιδεύει. Εγώ όμως θα ήθελα να αναφερθώ στην επικουρικότητα. Γιατί πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, θα μπορούσαν να το έχουν κάνει τα κράτη-μέλη, αλλά προφανώς δεν γίνεται. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Θεωρώ λοιπόν πως για λόγους δικαιωμάτων των πολιτών να, πως θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα κράτη-μέλη μόνα τους δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι τέτοιο προς το συμφέρον των πολιτών. Thank you very much. συνάδελφος Χάντλικ. ευχαριστώ. Μιλάμε όχι για έλλειψη ε, ρύθμισης, αλλά για έλλειψη εφαρμογής πάλι. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από όταν υιοθετήσαμε το σχετικό ψήφισμα, αλλά βλέπουμε πως πολλοί Ευρωπαίοι ακόμα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του 112 και όσοι το γνωρίζουν βλέπουν πως δεν λειτουργεί σωστά. Και ανταυτού μετά το, αντί για βοήθεια τους λένε πάρτε ξανά το τάδε νούμερο. Πότε λοιπόν θα ληφθούν ε, μέτρα, ειδικά για το αντίστροφο 112 για να ενημερώνουμε δηλαδή τους πολίτες μας ε, για μια φυσική καταστροφή η οποία θα πλησιάζει. Επίσης ε, είχαμε εγκρίνει το ψήφισμα για την οδική ασφάλεια και μιλήσαμε για το σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης στα αυτοκίνητα που θα έπαιρνε υποτίθεται το 112 και θα ενημέρωνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ατυχήματος για να υπάρχει γρήγορη αντίδραση αλλά πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα 112 πρώτα. Η Κομισιόν έχει οθετήσει τη σχετική πρόταση. Τι γίνεται όμως με την εφαρμογή, μπορεί να μας ενημερώσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, επί της αρχής ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό νούμερο είναι μια πρακτική λύση και ταυτόχρονα βέβαια θα μπορούσαν να καταργηθούν τα εθνικά νούμερα αλλά βλέπουμε εδώ πέρα πως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την σύνδεση των κλήσεων και θα έπρεπε νομίζω να υπάρχει μια παρόμοια ταχύτητα και επαγγελματισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι στοιχειώδες επίσης. Η Κομισιόν θα μπορούσε να ορίσει κάποιες προδιαγραφές με βάση το σβέλτιστες πρακτικές, όπως παραδείγματος χάρη αυτές οι οποίες υπάρχουν στην ε, Αυστρία. Και βεβαίως να οριστούν ε, κάποια κριτήρια αποτελεσματικότητας και μία προσέγγιση εξυπηρέτησης του πολίτη, να υπάρχουν επίσης και τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ε, απαιτήσει των πολιτών. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ομπερμάγερ και τελευταίος μιλητής στη διαδικασία του Catch the Eye, ο συνάδελφος Μπόρτς. E, e, Σας ευχαριστώ. Το θέμα του 112 είναι κάτι το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση την κοινή Ευρώπη. Σήμερα, τη σήμερα ημέρα, στην εποχή της κινητικότητας, η ασφάλεια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν πια συγκεκριμένα να εισαχθεί αυτή, αυτό το μέτρο και να παρακολουθηθεί το, η κατάσταση προόδου της εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Βέβαια λειτουργεί σε όλες τις χώρες, αλλά χρειάζεται καλύτερο συντονισμός και έπειτα χρειάζεται να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πολυγλωσία διότι Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα ατύχημα ε, μειώνονται από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερα στις ε, ε, συνοριακές περιοχές ε, πρέπει να υπάρχουν ε, τηλεφωνητές και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το νούμερο 112 δωρεάν για όλους όσους περνούν τα σύνορα. Ευχαριστώ. Up to Commissioner Και τώρα ο Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους βουλευτές για το συνεχές ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το νούμερο 112. Η Κομισιόν υπαγρυπνεί και στηρίζει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές να προωθήσουν το νούμερο αυτό. Θα συνεχίζουμε να ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο για τα, σχετικά με, το πώς προχωρούν τα θέματα που ε, θέσατε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να καλέσω τώρα εγώ εσάς να ενθαρρύνετε τις χώρες σας να προωθήσουν το νούμερο αυτό. Ευχαριστώ. Αδελφοί, η συζήτηση γύρω από την προφορική ερώτηση έληξε και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση της κυρίας Κάμερβερτ για τη συνδεδεμένη τηλεόραση και ήθελα να παρακαλέσω την ε, εισηγήτρια να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά.